Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω θερμά στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ολομελίας ε, και εκ μέρους όλων μας τον κύριο Ιγκόρ Κόρμαν που είναι πρόεδρος της ε, Μολδαβικής Βουλής και να καλωσορίσω και την αντιπροσωπεία του που έχει ε, εγκατασταθεί στο θεωρείο για να παρακολουθήσει τη συζήτηση για τη Μολδαβία και να γίνουν μάρτυρες της ιστορικής αυτής ψηφοφορίας για την έγκριση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Μάλιστα, η αντιπροσωπή αυτή από τη Μολδαβία θα συναντήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλές αντιπροσωπείες και επιτροπές του Κοινοβουλίου μας. Εκ μέρους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου σας εύχομαι θερμά, λοιπόν, θα σας